Αγαπητοί συνάδελφοι, αν είμαστε έτοιμοι, να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Και συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Συνεπώς, έτοιμοι όλοι. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα κάνουμε, έτσι. Πρόκειται για την έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή τη οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα υποστήριξη και προστασία θυμάτων εγκληματικότητα. Έτοιμοι όλοι. Η Αντζέλικα Μολινάρα και η Τερέσα Χιμένε Μπεθερίλ Μπάριο είναι οι συνεισηγήτριε. Δεν ξέρω πριν την ψηφοφορία μήπω θέλετε να πείτε κάτι. Τερέσα, δύο λόγια μόνο, ε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδες εισηγητές για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Στην έκθεση αυτή εννοείται όλοι θέλουμε να υποστηρίξουμε τα θύματα, παντός είδους θύματα εγκληματικότητας είδαμε ότι υπάρχουν χώρες που ακόμα δεν εφαρμόζουν σωστά την έκθεση του 2012 που εκπονήσαμε. Οπότε θέλουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις αδυναμίες, να υπάρχει περισσότερη κατάρτιση για την αστυνομία, περισσότερη ενημέρωση για το κόσμο, καλύτερη εκτίμηση ε, της κατάστασης για κάθε θύμα, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες κάθε θύματος που μπορεί να είναι ευάλωτο, είτε είναι παιδί, γυναίκα, άτομο με αναπηρίες, οτιδήποτε από οποιοδήποτε οργανωμένο έγκλημα και προσθέσαμε, γιατί τότε δεν είχαμε τόσες ε, επιθέσεις το 12, συμπεριλάβαμε και κάτι για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των θυμάτων τρομοκρατίας ε, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους τους και ηγητές, τη γραμματεία, τις πολιτικές ομάδες που μας ε, βοήθησαν, τους βοηθούς όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είσαστε εδώ παρόντες όλοι για να στηρίξετε αυτή την υπόθεση, για να προστατεύσουμε τα θύματα εγκληματικότητας ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μολινάρ. Εσείς μήπως. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Εκ μέρου τη Επιτροπή Γυναικών θέλω να ευχαριστήσω όλου του σκιώδει εισηγητέ. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνεισηγήτρια από την ΛΥΜΠΕ η συνεργασία μας, θέλω να το τονίσω αυτό, ήταν απόλυτα καρποφόρα. Ίσως οφείλεται σε αυτό ότι ήμασταν ουσιαστικά αποκλειστικά γυναίκες που συνεργαστήκαμε για αυτή την υπόθεση. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία. Σήμερα στην ψηφοφορία ελπίζω να πετύχουμε ευρεία συνένεση και επειδή οι γυναίκες θύματα έχουν μια διαφορετική εμπειρία από τα θύματα άντρες στην κοινωνία μας. Αυτό αντικατοπτρίζεται πολύ καλά στην έκθεση, οπότε ελπίζω να έχουμε ευρεία στήριξη. Πρόεδρος, ωραία. Ακούσαμε τις δύο συνηγήτριες από τις δύο επιτροπές. Η κυρία Μπλεκεβουτσίτε και εγώ, εννοείται, ευχαριστούμε επίσης όλους σας. Περνάμε στην ψηφοφορία, αλλά να πω προηγουμένως ότι η κυρία Σίλστρα αποσύρει το όνομά της από την τροπολογία 75. Οπότε ψηφίζουμε πρώτα τροπολογία 78. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 79. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 80. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 8. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 10. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 100. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 101. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 12, λέει ο Πρόεδρος. Α, συγγνώμη. Συμβαστική 11 πρώτα. Συμβαστική 11 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. 11, ναι, συγγνώμη. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τώρα συμβαστική 12. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 114. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 124. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 13. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Νομίζω ότι από τους πράσινους και την ΚΟΕ ψηφίζουν ένας παραπάνω κάθε φορά. Μια στιγμή, συνάδελφοι. Εντάξει, συγγνώμη, ένα τεχνικό ζήτημα ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τροπολογία 136. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε για την 136 παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 14. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 15. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 120. Ψηφίστε. Τέλος. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε την 120. 120 λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος της προφορίας. Απορρίφθηκε. Πρέπει να κλείσουμε και να ξανανοίξουμε τα μηχανήματα γιατί κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει. Οπότε, αν δεν λειτουργεί, πηγαίνετε σε ένα άλλο μηχάνημα. Ή αλλιώ δυνατά του χειρό εσεί και θα, υπολογίζουμε, θα συνυπολογίζουμε την ψήφο σα. Λοιπόν, ξαναβάζουμε τα μηχανήματα να δουλέψουν. Επανεκκίνηση του μηχανισμού. στο μηχάνημα που δείχνει την ψηφοφορία των μελών της Επιτροπής Γυναικών φαινόταν ένας παραπάνω να ψηφίζει, ενώ στο άλλο μηχάνημα όχι. Πραγματικά τεχνικό το ζήτημα. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, όχι. Η Λίμπε έχει κακή φήμη. Καθαρά τεχνικό το ζήτημα, έτσι δεν είναι. κίνηση των μηχανημάτων. Και είναι σημαντικό για την τελική ψηφοφορία, όπως καταλαβαίνετε. Συνάδελφοι, Να το κάνουμε παλιωμοδίτικα, δυνατά της χειρός. Ωραία. Τροπολογία 123 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 155 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω να το λέξουμε. Μπορούμε. Δεν μπορούμε. Ξανά λοιπόν, για να δάσω στις χειρός θα μετρήσουμε καλύτερα. Υπέρ, κατά, εντάξει, εγκρίνεται. Τροπολογία 156 υπέρ, κατά, αποχές, εδώ ήταν πιο δύσκολα. Λοιπόν, εσείς που είσαστε αντιπρόεδρος έχετε τη συνήθεια ίσως. Ωραία, ξαναψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι λέτε. Πώς θα το ελέγξουμε. Γι' αυτό είναι πάντα καλύτερα να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Είμαστε έτοιμοι. Εγκρίνεται. 156 θα μετρήσουμε. Λοιπόν, ξαναψηφίστε χέρια και μετράμε. Υπέρ. «22 υπέρ, κατά, 24 υπέρ 22 κατά. Εγκρίθηκε. 121 τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 160 με προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Αποχές. 159 τώρα. Α, καταπίπτει. Συμβαστική 19, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 180 και 181 είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 193 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ, α όχι καταπίπτει. 195 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 198 τώρα. Α, θέλετε να ελέγξουμε για την 195. Ωραία. Ελέγχουμε υπέρ. Ηλεκτρονικά δεν μπορούμε, οπότε δυνατά στους χειρός. Σηκώστε τα χέρια σας καλά και κρατήστε τα 195 λοιπόν υπέρ. Μετράμε. 23 κατά. 18 κατά. Αποχές. Ωραία, εγκρίθηκε. 196 κατά 198 <coughs> υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ κατά αποχές. Θα μετρήσουμε. Λυπάμαι. Λοιπόν, υπέρ. Κρατήστε τα χέρια σας. Ανεβασμένα. Α, εγκρίθηκε, εντάξει. 204 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 218 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 219 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται 223 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται 226 υπέρ, όχι κατά αυτή, 227 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 228 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική. Α, τώρα έχουμε η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ε? σωστά. Λοιπόν, συμβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να συνεχίσουμε έτσι. Ωραία, θα έχουμε μόνο. 234 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. 245. 239, να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 239. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 21-17. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 247 αλλά καταπίπτει. 246 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανείς δεν σκόνει χέρια. Επειδή ξέρετε δηλαδή ότι δουλεύει το μηχάνημα τώρα, τα τεμπελιάζετε. Ωραία. 246 ηλεκτρονικά λοιπόν, ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 248, ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Αναφορές. Αριθμός 1. ε, ψηφίστε μάλλον ηλεκτρονικά. Τέλος, εγκρίθηκε. 2. Ψηφίστε. Τέλος, εγκρίθηκε. 3. Ψηφίστε. Τέλος, εγκρίθηκε. 4. Ψηφίστε. Τέλος, εγκρίθηκε. 5. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 6. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 7. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε να τις ψηφίσουμε μαζί. 8 με 13. 8 μέχρι και 13. Ψηφίστε παρακαλώ μαζί όχι, όχι, υπάρχει μια αντίρρηση σε αυτό. Όχι τότε. Λοιπόν, 8. Ε, στην 8 είμαστε. 8. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 8 αναφορά. Τέλος, εγκρίθηκε. 9. Ψηφίστε. Τέλος, εγκρίθηκε. 10. Ψηφίστε. Τέλος, εγκρίθηκε. 11. Ψηφίστε. Τέλος, εγκρίθηκε. 12 ψηφίστε. Τέλος εγκρίθηκε. 13 ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 14 και 15 είναι ίδιες. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος εγκρίθηκαν. 16 και 17 είναι ίδιες. Ψηφίζουμε. Τέλος εγκρίθηκαν. 18 και 19 είναι ίδιες. Ψηφίζουμε. Τέλος 18 και 19 είναι ίδιες. Ψηφίστε. Ξανά. Ωραία, 18 και 19. Ξανά. Ψηφίζουμε 18 και 19. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. 20. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε 21. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 22. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 23. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. 24. Εγκρίθηκε 23. 24 λοιπόν ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 24. Ναι. Τώρα 24. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική αριθμό 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 29. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 30. Ψηφίστε. Τέλος. Πιο αργά να πηγαίνω, λέτε. Καλά, θα πηγαίνω λίγο πιο αργά. 30 λοιπόν, εντάξει, ψηφίσατε, εγκρίθηκε. 31. Με προφορική, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 32. Μπορείτε να ψηφίσετε. 32. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Πιο αργά είπατε. Πάω πιο αργά. Και το μηχάνημα πάει αργά. Ναι, ναι, κλείνει η ψηφοφορία. Λοιπόν, συνάδελφοι, 33. Ξανά. Ψηφίζουμε ξανά 33 ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 34. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 3. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 40 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 42. Ψηφίστε. Τέλος. 42. Ψηφίστε. Α, την κάναμε αυτή. 44 ήμασταν. Ωραία. Ψηφίστε. 44. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 45. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 47. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 49. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 50. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 4. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 5. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 53 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 54. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 55. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 56. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 6 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 65. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 69. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 66 και 71 που είναι ίδιες. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 73 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 74. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 75 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 76. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 77. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε και αυτή. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε 42 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια και στις δύο συγγήτριες. Thank you, colleagues, for your patience. I'm sorry. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, αγαπητοί συνάδελφοι.